στον Μπουρούντι. Ο κύριος Νέβεν Μίμητσα εκπροσωπεί την κυρία Μογκερίνη και του δίνω αμέσως με χαρά το λόγο παρακαλώ κύριε Επίτροπε. Thank you very much, Mr. President. Honorable... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, είμαι μέλη του Κοινοβουλίου. Χαίρομαι που μου δίνεται αυτή η ευκαιρία να απευθυνθώ στο Κοινοβούλιο, το οποίο μέσω των προηγουμένων ψηφισμάτων του και δράσεων του έχει υπενθυμίσει στο λαό του Μπουρούντι ότι τον υποστηρίζει στην προσπάθειά του να βρεθεί μια διέξοδος στη βιώση και να αποκτήσει μια βιώσιμη δημοκρατία με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με ανάπτυξη και να καταφέρει να υπάρξει περιφερειακή ένταξη του Μπουρούντι στην περιοχή του. Ωστόσο, τα σημαντικά επιτεύγματα των Μπουρούντι των τελευταίων ετών αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κίνδυνο. Εξαιτία τη απόφαση του κυβερνώντος κόμματος να ορίσει τον πρόεδρο Νκουρουζίζα ως τον υποψήφιό του για τρίτη συνεχόμενη θητεία που έχει δημιουργήσει μεγάλες ανατερεχές στο εσωτερικό της χώρας. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί αμέσως. Στα ε, συμπεράσματα του, Μαΐου, του Μαρτίου του Συμβουλίου ε, των Υπουργών Εξωτερικών ε, τονίστηκε η σημασία της Συμφωνίας της Αρούσα και την ανάγκη που υπάρχει ε, να βρεθεί μια λύση που στη βάση αυτής της ε, συμφωνίας. Ιδιαίτερα όσον αφορά το ζήτημα της τρίτης θητείας του Προέδρου. Αυτή παραμένει η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ακόμα χρόνος για να βρεθεί διέξοδος μέσω διαλόγου και συμφιλίωσης. Η ύπατη εκπρόσωπος Μογκερίνη είναι ιδιαίτερα ανήσυχη εξαιτία των αναφορών που λαμβάνουμε για συλλήψεις ε, ε, δημοσιογράφων, μελών της κοινωνίας των πολιτών, για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για αστυνομική βία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε υποστηρίξει την ε, απελευθέρωση του ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήδη πέρυσι. Έχουμε ήδη λάβει αναφορές ότι έχει επανασυλληφθεί χωρίς κάποια αιτιολόγηση. Χαίρομαι που αφέθηκε ελεύθερος και συγχαίρω εκείνους που έχουν προσπαθήσει να, για αυτή την απελευθέρωση του. Ωστόσο, ο, του κυρίου Μπονίμπα. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίοι κινδυνεύουν και αυτούς θα πρέπει να τους υποστηρίξουμε. Η παρενόχληση των απερασπιστών ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοσιογράφων και οποιοδήποτε ασκή κρατική πρέπει να σταματήσει. Κύριε Πρόεδρε, Θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες εκείνων που ε, δολοφονήθηκαν ή ε, τραυματίστηκαν στις πρόσφατες αναταραχές. Καθώς ε, επίσης να εκφράσω την ανησυχία μου για τι περιορισμού που επιβλήθηκαν στα μέσα μαζική ανεμέρωση και στο δικαίωμα του συνεθρίζεστε. Κάτι που δεν δίνει τη δυνατότητα στους, ε, στο λαό του Μπουρούντι να καταλάβει τι συμβαίνει, ιδίω σε μια προεκλογική περίοδο. Κάτι που οξύνει τα πάθη και οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερε και εντονότερε συγκρούσει στου δρόμου. Είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή να επικρατήσει η λογική, να μην υπάρχουν προκλήσεις κατέρωθεν οι αρχές του Μπουρούντι να προσπίσουν το δικαίωμα στην ελευθερία της ε, συνάθρησης και να μην ε, επιτρέπουν την υπερβολική χρήση βίας από τις αστυνομικές αρχές. Όσον αφορά τώρα τις ε, προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στο Μπουρούντι, έχω να δηλώσω τα εξής. Όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει οικονομική βοήθεια στις, ε, για την διοργάνωση των εκλογών και επίσης θα αποστείλει παρατηρητές. Αυτό είναι μια σημαντική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δείχνει ότι είμαστε αποφασισμένοι να είναι επιτυχείς αυτές οι εκλογές. Ωστόσο, στην ε, πρόσφατη δήλωση της, ε, κυρίας, της εκπροσώπου της κυρίας Μογκερίνη αναφέρεται επιλέξει ότι η παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η παρενόχληση, οι απειλέ. και οι δολοφονίε είναι στοιχεία που θα πρέπει να αποφευθούν, να λείπουν τελείω από μια προεκλογική περίοδο και θέλω να το επιθυμίσω αυτό στις ε, αρχές του Μπουρούντι. Στι 13 Απριλίου απίφθηνε επιστολή η κυρία Μογγερίνη στη βάση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του Μαρτίου, υπενθυμίζοντα στι αρχέ του Μπουρούντι ότι όλοι οι πολιτικοί ε, παράγοντες, όλοι οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην εκλογική διαδικασία και επίσης να υπάρξει πλήρης πρόσβαση στους παρατηρητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Σύμφωνα με τη Συμφωνία του Κοτονού, είναι ξεκάθαρο ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία. Ο σεβασμό για το ανθρώπινο δικαίωμα και το κράτο δικαίου αποτελεί θεμελιώδε στοιχείο αυτή τη συμφωνία. Επομένω, δεν θα ανεχθούμε παραβιάσει τέτοιε. Και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υπόλοιποι διεθνεί παράγοντε θα πρέπει να προσπαθήσουν να προωθήσουν το διάλογο, να βοηθήσουν να υπάρξει κάποια συμφωνία ή κάποια συνένεση ανάμεσα στους διάφορους πολιτικούς ε, του Μπουρούντι και την κοινωνία των πολιτών στο Μπουρούντι. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε όλες τις ε, δυνατότητες που έχουμε στη διάθεσή μας, αναλύουμε τις επιπτώσεις που θα έχει η σημερινή κατάσταση με, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και επίσης εξετάζουμε την ανάληψη δράσης επί τη βάση της Συμφωνίας του Κοτονού. Έχοντας λοιπόν αυτά υπόψη, θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι οι υπεύθυνοι των αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν, σύμφωνα και με το άρθρο 8 της Συμφωνίας του Κουτονού, εντείνει τις επαφές τους με τις αρχές του Μπουρούντι. Όταν μιλώ για πιθανά μέτρα ωστόσο, θέλω να είμαι ξεκάθαρος ως προς το εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους σημαντικότερους εταίρους της αναπτυξιακής συνεργασίας με τον Μπουρούντι και θα θέλαμε να δώσουμε τη δυνατότητα να αποφευχθεί μια επιδείνωση της κατάστασης ε, στην χώρα αυτή η οποία θα είχε δυσμενείς συνέπειες για μεγάλα μέρη του πληθυσμού της. Και αυτό είναι η κατευθυντήριά μας ε, ε, αρχή με βάση της οποία, στην οποία διπλασιάσαμε την αναπτυξιακή βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς το ε, Μπουρούντι από και έφτασε τα 432 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αναζητούμε λύσεις θετικού χαρακτήρα που θα επιτρέψουν στο λαό του Μπουρούντι να εκπληρώσει τις προσδοκίες του. Πρέπει να φροντίσουμε η όποια δράση λάβουμε να μην έχει δυσμενές αντικτυπώσεις στους στοχούς και οι σχέσεις με τον Μπουρούντι να αποκατασταθούν και να εξομαλυνθούν όσο το γρηγορότερο γίνεται. Ως Επίτροπος Αρμόδιος για την ε, Αναπτυξιακή Συνεργασία πρέπει να ε, τονίσω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ιδιαίτερα και να καταπολεμήσουμε τη, χρήση των ε, χρηματοδότησης της αναπτυξιακής ε, συνεργασίας για ε, καταπίεση. Ευχαριστώ. Και τώρα ακολουθούν οι πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για 1,5 λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Γιώχη Μτσέλα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, Σήμερα το πρωί εδώ μιλήσαμε για τους πρόσφυγες που ψάχνουν σωτηρία στην Ευρώπη και ακούστηκαν φωνές που λένε ότι δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε μόνο τα συμπτώματα αλλά και τα αίτια αυτή τη κατάσταση στι χώρε καταγωγή των ανθρώπων αυτών που φεύγουν από την πατρίδα του. Γι' αυτό είναι σωστό και σημαντικό να ασχοληθούμε σήμερα με την κατάσταση στο Μπουρούντι, όπου τι τελευταίε ημέρε ο στρατό, αστυνομία και πολιτικέ ομάδε αντίπαλε ε, ε, ε, προβαίνουν σε βιοπραγίε. Έχουμε και νεκρού. 10.000 είναι ήδη πρόσφυγε και σε γειτονικά κράτη. Οπότε η σύγκρουση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στο Μπουρούντι. Μετά από δεκαετίες εμφυλίων πολέμων και εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και πρόσφυγες ήταν στο παραπέντε μιας δημοκρατικής δοκιμασίας ε, τον ε, Μάιο ε, βουλευτικές εκλογές και τον Ιούνιο προεδρικές. Ο νυν πρόεδρος Νούρουν Κουζίζα αντισυνταγματικά δήλωσε ότι θέλει να είναι υποψήφιος για τρίτη θητεία ε, που δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα και αυτός φταίει για τη σημερινή κατάσταση. Η διεθνής κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ασκήσει πίεση στους ηθήνοντες εκεί για να αποφευθεί μια νέα ανθρώπινη κατάσταση καταστροφή και τραγωδία στη χώρα. Το είπε και ο Επίτροπος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την παραγω... ε... αποστολή παρατήρησης των εκλογών θα πρέπει να δείξει ότι παρακολουθεί την κατάσταση και δεν τη είναι καθόλου αδιάφορη η κατάσταση στη αφρικανική αυτή χώρα. Ευχαριστώ κύριε Τσέρ. Ο κύριος Πιτέλα τώρα, πρόεδρος της ε, ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πίτροπε, το κλίμα της ε, βίας, του τρόμου, του εκφυβισμού που οθεί χιλιάδες ανθρώπους προς τη Ρουάντα, τους τρέπει σε φυγή, ε, δίνει την ε, δυνατότητα να ξεσπάσει νέα εθνική σύρεξη στο Μπουρούντι και μας ανησυχεί. Ε, και ο απερχόμενος πρόεδρος επέλεξε να θέσει υποψηφιότητα για μια θητεία παραβίαση τη συμφωνία τη Ρούσια και αυτό κινδυνεύει να οθήσει τον Μπουρούντι σε ένα παρελθόν εθνικής βίας θυμάται τη διαδικασία δημοκρατισμού της χώρας. Πριν λίγες εβδομάδες, ε, εγώ μαζί με μία αποστολή της ομάδας μου επισκέφθηκα τον Μπουρούντι και την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών οι λόγοι της γενοκτονίας του 1994 εξακολουθούν να υπάρχουν εκεί. Απλώς είναι υπόγειοι. Εμείς δεν μπορούμε με διαφορία να αναμένουμε ε, να γεννηθεί ένα νέο τέρας. Πρέπει να δράσουμε αμέσως. Γνωρίζουμε ότι είπατε εκπρόσωπος παρακολουθεί εκ του συνεγγύς και με αποτελεσματικότητα την εξέλιξη της κατάστασης και της απευθύνουμε έκκληση για να ασκήσει πίεση στον πρόεδρο να μην θέσει εκ νέου Όμω, εγώ απευθύνω και άμεση έκκληση στον πρόεδρο θέλετε κύριε πρόεδρε του Μπουρούντι ε, να αγκυλωθείτε σε μια εξουσία ε, χωρίς λαό ή θέλετε να γίνετε ένας καθοριστικός παράγοντας ε, στην δημοκρατική μετάβαση της χώρας σας κύριε πρόεδρε σκεφτείτε το εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά θα κάνουμε αυτό που μας αναλογεί ε, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πιτέλα. Και τώρα από τους συντηρητικούς για 1,5 λεπτό κυρία Άννα Φωτίγκα. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Το Μπουρούντι βρίσκεται σε μία από τις ε, πιο ασταθείς ε, και πιο φτωχές περιοχές του κόσμου. Μιλούμε για την ευρύτερη περιοχή των μεγαλών λιμνών ε, και ξέρουμε ότι έχουμε εμφυλίους πολέμους στην ευρύτερη περιοχή και ήδη Έχουμε δει τέτοια παραδείγματα στη Ρουάντα και στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό και γνωρίζουμε ότι οι ειρηνευτικέ συμφωνίες που υπογράφτηκαν στην Αρούσα είναι ιδιαίτερα εύθραστες. Όμως ε, οδήγησαν στο να έχουμε μεγάλες προσδοκίες και φυσικά θα θέλαμε να δούμε ε, να Έχουμε καλές εξελίξεις στη χώρα όμως. Ε, αποφασίστηκε από το κυβερνών κόμμα να ε, ανακοινώσει την θητεία του σημερινού Προέδρου για τις προεδρικές εκλογές για τρίτη φορά και αυτό, την υποψηφιότητα με συγχωρείτε, και αυτό φυσικά παραβιάζει τις συμφωνίες ε, της Αρδούσα και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα κύρια στοιχεία που οδήγησαν στο ξέσπασμα διαμαρτυριών στη χώρα γιατί φυσικά υπενθυμίζει την ε, τρομακτική περίοδο του εμφυλίου πολέμου και γνωρίζουμε ότι η ύπατη εκπρόσωπος, η κυρία Μαγκερίνη, μπορεί να βασιστεί στην ε, υποστήριξη της δικής μου πολιτικής ομάδας για οποιαδήποτε προσπάθεια καταβάλει για να προσπαθήσει να εγγυθεί την ειρήνη στο Βουρούντι. Γιατί προφανώς πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η όλη εκλογική διαδικασία θα είναι δίκαιη και θα διέπεται από Και για να το πράξουμε αυτό, χρειαζόμαστε αποστολή παρατήρηση των εκλογών. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι εκλογέ θα λάβουν χώρα σε δημοκρατικό πλαίσιο και νομίζω ότι θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα δημοκρατικά τεστ για τη χώρα. Ευχαριστώ για δύο λεπτά από του φιλελευθέρου, κύριε Χέλντε Βάουτμαντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, υποψηφιότητα του απερχομένου Προέδρου για τρίτη θητεία ε, άναψε φυτίλια. Και αυτή είναι η κατάσταση σήμερα στο Μπουρούντι. Καταλαβαίνουμε τι επίκρατη ε, στην ε, περιοχή. Είναι μπαρουταποθήκη με πολλές ζώνες συγκρούσεων και μια ειρήνη στο Μπουρούντι που είναι πάρα πολύ εύθραυση και τώρα δοκιμάζεται. Στην Ευρώπη έχουν γίνει λάθη από διάφορα κράτη-μέλη. Πολύ συχνά Κλείσαμε τα μάτια και είπαμε καλά, είναι βία στην Αφρική εκεί πέρα, σκοτώνονται. Τώρα όμως έχουμε την ευκαιρία ε, να αποφύγουμε μια επατοχυσία. Και χωρίς ταμπού θα πρέπει να μιλάμε για μια γενοκτονία που προετοιμάζεται και επίκειται. Έχω επισκεφτεί προσωπικά τη Ρουάντα μετά τη γενοκτονία του 1994 και πρέπει να σας πω ότι είδα φρικτά πράγματα. Ε, καινοτάφια, ε, ε ομαδικούς τάφους, ε, κρανία, ανθρώπινα μέλη, άνδρες, γυναίκες, παιδιά που είχαν ε, θανατωθεί και μόνο που το θυμάμαι ανατριχιάζω ότι κινδυνεύει κάτι τέτοιο να επαναληφθεί στο Μπουρούντι. Σήμερα δεν θέλουμε μόνο συζήτηση, χρειαζόμαστε και έργα το θέμα δεν είναι να στέλνουμε συλληπιτήρια σε οικογένειες και να ζητάμε συγγνώμη. Τι να τις κάνουν τις ε, συγγνώμες και τα συλληπιτήρια οι άνθρωποι. Δεν γυρίζουν πίσω οι νεκροί τους. Χρειάζεται υποστήριξη λοιπόν από όλες τις πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ομιλήτρια από την ΚΟΗ, κυρία Βαζιά, για μισή λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το 2000 συμφωνίες της Αρούσα τερμάτισαν ε, χρόνια ε, εμφυλίου πολέμου στην, στο Βορούντι μεταξύ Χούτου και Τούτσι. Και ε, ο πρώτος πρόεδρος Χούτου στην ιστορία της χώρας εξελέγει. συμφιλίωση και νέο σύνταγμα ακολούθησαν. Και ε, η απόφαση του απερχομένου Προέδρου να διεκδικήσει και τρίτη θητεία διακυβεύει την εύθραυστη ισορροπία. Εδώ και εβδομάδες ε, ακούμε ότι πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Ακολούθησε η απόφαση του συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος ε, διαμαρτυρίες και μαζική καταστολή. Ήδη οι ΜΚΟ μετρούν θανάτους και εκατοντάδες συλλήψεις. Τα μέλη του κόμματος ε, στην εξουσία πρωτοστατούν στις βιοπραγίες ε, και ε, στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος όπως πρόσωπος του Προέδρου και του κόμματος ε, έχουν καθαιρεθεί. Πάνω από 20.000 ε, άνθρωποι έχουν φύγει από τη χώρα γιατί φοβούνται για την ασφάλεια και την ακαιρεότητά τους. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσει τις αρχές και τον πρόεδρο της χώρας και αν χρειαστεί να ε, συνδέσει τη βοήθεια της, την οικονομική της Ένωσης γιατί η χώρα εξαρτάται για 50 και πλέον από την εξωτερική βοήθεια. Θα πρέπει οι εκλογές να είναι δίκαιες και διαφανείς. Γνωρίζουμε ότι ότι η φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ακούγονται στον Μπορούντι. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε αυτή την περιοχή να αποσταθεροποιηθεί ακόμα περισσότερο. Χρειάζεται ταχεία δράση για να αποφευθεί νέα αιματοχυσία. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ομιλήτρια, η Μαρία Χόιμπουχ, για 1,5 λεπτό από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, σωστά περιγράψατε την κατάσταση στον Μπορούντι, ε, καταδείξατε τα προβλήματα και είπατε και πόσο εύθραυστη είναι η κατάσταση εκεί. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τα όσα λέτε, ε, υποθέτω ότι είναι πολύ ε, κριτική η ματιά σας και για την αντιπολίτευση. Είναι ανίποτα αυτά που συμβαίνουν εκεί. Και σας ερωτώ, μιλήσατε για αποστολή παρατήρησης των εκλογών, από ποιους θα απαρτίζεται, θα είναι υψηλόβαθμα, στελέχη, ποιοι θα πάνε εκεί, είναι πολύ σημαντικό για να δώσουμε, ε, στείλουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση. Επόμενη ερώτηση. Ποια μέτρα λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για καλό συντονισμό και συνεργασία με όλες τις υπόλοιπες διεθνείς ε, παρατήρησης των εκλογών και χρειάστηκε υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών εκεί. Το έχετε σκεφτεί να τη συμπεριλάβετε εκ των υστέρων μετά τις εκλογές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει ε, τι θα κάνει με τη μακροοικονομική βοήθεια που δίνουμε εκεί. Αν επανεκλεγεί ο πρόεδρος θα το παγώσουμε αυτό. Πρέπει να το συζητήσουμε και δημόσια και να λέμε τις προθέσεις μας. Διότι έχουμε εδώ ένα μέσο για να ασκήσουμε πίεση σε αυτό τον πρόεδρο και όχι μόνο με λόγια αλλά και με έργα. Και σε περίπτωση που δεν προτίθεστε να τα παγώσετε αυτά, πώς θα εξασφαλίσετε ότι ε, τα χρήματα θα πηγαίνουν στους πραγματικούς δικαιούχους, δηλαδή στον πληθυσμό και στο λαό και όχι σε τσέπες της κυβέρνησης για αλότριους σκοπούς. Υπάρχει το άρθρο 96 της Συμφωνίας Κοτονού που μιλάει για ε, ε, δυνατότητα αναστολή των σχέσεων μας με το Βουρούντι. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό η κυρία Κασέτου Κενγκέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα βρισκόμαστε ενώπιον μιας μεγάλης ευθύνης από την οποία δεν μπορούμε να διαφύγουμε. Βλέπουμε μια σφαγή που μπορεί να λάβει στην Κεντρική Αφρική διαστάσεις γενοκτονίας. Ναι, γενοκτονία. Πολύ συχνά το να μην αναφέρουμε, να μην προφέρουμε αυτή τη λέξη μας οδήγησε στο να παρατηρούμε ε, το μακελιό αθών. η υποψηφιότητα του Προέδρου Κρουσίζα για τρίτη θητεία είχε ε, αρνητικές συνέπειες στον Περουντό. Εμείς ε, καταγγέλουμε την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, τον περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας του τύπου που υλοποιεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Εγώ θα ήθελα ε, να ανοίξουν και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που έκλεισαν αρχικά το RPA. Εμείς, αν είναι δυνατόν, θα θέλαμε να ε, χρησιμοποιήσουμε και τη δυνατότητα μεμονωμένων επιβολής, μεμονωμένων κυρώσεων. Ε, ο φίλιος πόλεμος, ο Μπουρούντι, στο παρελθόν επεκτάθηκε στη Ρουάντα και προκάλεσε μία από τις πιο ντροπιαστικές σφαγές στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τώρα δεν μπορούμε πλέον πάλι να πούμε ότι είμαστε δύναμη για να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια του επικεφαλής της αποστολής ε, του ΙΕ στη Ρουάντα κατά τη γενοκτονία. Ε, ουσιαστικά αυτό που θα κάνουμε θα είναι να σφιξούμε το χέρι του διαβόλου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό η κυρία Μακάβα. Um, thank you, Mr. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας καλωσορίζω την ε, δήλωσή σας και τη δήλωση της σε προσώπου. Πρέπει να τερματιστεί η βία τώρα η αστυνομική βία, οι μαζικές συλλήψεις, ε, η καταπίεση των αντιφρονούντων, της αντιπολίτευσης, των ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όλα αυτά είναι ανεπίτρεπτα σε μια προεκλογική περίοδο και πρέπει να σταματήσουν τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη να υποστηρίξει το Μπουρούντι και να δημιουργηθεί μια, ένα βήμα για να, έτσι ώστε να γίνεται ένας ειρηνικός διάλογος που θα οδηγήσει σε ειρηνικές εκλογές. Οι εκλογέ αυτέ, όπω είπατε και εσεί, έχουν εξαιρετική σημασία όχι μόνο για τον Μπουρούντι, αλλά για ολόκληρη την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, μια περιοχή στην οποία στου επόμενου 18 μήνε θα υπάρξουν και πολλέ άλλε εκλογέ. Επίτροπε, το είπε, είπατε ότι έχουμε αυξήσει την αναπτυξιακή μα συνεργασία προ τον Μπουρούντι. Είμαι πρόεδρο τη Επιτροπή τη Αναπτυξιακή Συνεργασία και θα ήθελα να δω η αναπτυξιακή μας βοήθεια να πηγαίνει προς το σωστό σκοπό, δηλαδή να βοηθάει τους ανθρώπους επιτόπου τις υπηρεσίες που τους παρέχονται. Και αυτό είναι αδύνατο εάν δεν υπάρχει ειρήνη και σταθερότητα. Γι' αυτό η κυβέρνηση του Μπουρούντι πρέπει να εισακούσει τις ε, εκκλήσεις που τις απευθύνουμε. Βλέπουμε ήδη χιλιάδες ανθρώπους να περνούν τα σύνορα προς την ε, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, προς τη Ρουάντα. και φαντάζομαι θα συνεργαστείτε και με τον Επίτροπο Στυλιανίδη για να υπάρξει μια συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη για αυτούς τους πρόσφυγες. Κινδυνεύουμε αυτή τη στιγμή να γκριμιστούν όλα αυτά που χτίστηκαν τα τελευταία 15-20 χρόνια, γι' αυτό θα πρέπει να εξοκουστούν οι εκκλήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να ανακτήσει την δύναμη τη αυτή η χώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Λίντα για 1,5 λεπτό, Ελένα Βαλενθιάνο. Από το 2011 στο Μπουρούντι οι δυνατότητε ε, δημοκρατικής και πολιτικής συμμετοχή ε, σιγά σιγά το κυβερνόν κόμμα ε, και ο πρόεδρος εκφόβησαν και παρενόχλησαν τους πολίτες όμως η ανακοίνωση του πρόεδρου Κουρουσίσα για την απόφαση της υποψηφιότητά του επιδίνωσε τα πράγματα. Αυτή η απόφαση να παρουσιαστεί για μια τρίτη θητεία. Όπω είπαν οι συνάδελφοι και ο ίδιο επίτροπο, ε, θίγει ε, τι ειρηνευτικέ συμφωνίε τη και το πνεύμα του συντάγματος σε μια χώρα με ένα τόσο δραματικό παρελθόν και σε μια περιοχή με τόσο ε, εύθραστη σταθερότητα η απόφαση του Πρόεδρου Κουρουζίζα θέτει πολύ μεγάλο κίνδυνο για όλους. Είναι πολύ εύκολο, πρέπει να ζητήσουμε από τον Πρόεδρο να αναθεωρήσει την απόφασή του, πρέπει να ζητήσουμε από την κυβέρνηση να ξανανοίξει τους χώρους συμμετοχής στην πολιτική, τα ραδιόφωνα που έκλεισε, να απελευθερώσει τους πολιτικούς κρατουμένους ε, και να επιτρέψει τη δημοκρατική συμμετοχή και αν δεν είναι έτσι, κύριε Επιτροπέ, αν ο κύριος Πρόεδρος ε, δεν αλλάξει γνώμη και αν ε, δώσει τις θεμελιώδεις και πολιτικές ελευθερίες που είναι απαραίτητες για την εκλογική διαδικασία, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να υποστηρίξουν την εκλογική διαδικασία στον Μπορούντι, γιατί θα είναι ψευδής πλαστή και γιατί ο Κουρουζίσα θα χρειαστεί πολύ κατασταλή ε, για να υλοποιήσει αυτή την εκστρατεία. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε. Και τώρα ερχόμαστε στη διαδικασία κάτσιαί. Πρώτος ομιλητής για ένα λεπτό είναι ο κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ήδη έχω πάρει το λόγο για την κατάσταση του Μπουρούντε. Από είδαμε στην περίπτωση του κυρίου Νουγκουρίκα, ο οποίος ήταν δημοσιογράφος από το ραδιόφωνο Public African τώρα, ε, όσα συμβαίνουν ε, στις 25 Απριλίου, η σύγκρουση των πολιτών με τους αστυνομικούς είναι πιο σκληρές από την εποχή του Φιλίου Πολέμου. Ιδίως επλήγησαν τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες 48 ώρες ε, ε, διακόπησε είτε πλήρωση το μερικός ε, η διάδοση και συνελήφθησαν κάποιοι από τους δημοσιογράφους αφού ο πρόεδρος αφού επιτέλεσε δύο θητείες αποφάσισε να θέσει υποψηφιότητα για μία τρίτη θητεία καταπεραβιάζοντας το άρθρο 97 του συντάγματος. Θα πρέπει και η Ευρώπη αποφασιστικά να παρέμβει έτσι ώστε να βρεθούν δημοκρατικοί τρόποι διακυβέρνησης για να μην έχουμε νέο εμφύλιο πόλεμο στη χώρα και να εγγυθούμε και την ελευθερία της έκφρασης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάς για ένα λεπτό παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση στο Μπουρούντι μας απασχολεί άλλη μια φορά. Πριν από λίγο διάστημα είχαμε συζητήσει το θέμα αυτό, είχα τοποθετηθεί και για τις διώξεις που γίνονται κατά του δημοσιογράφου Νουκουρίκα. Είχαμε πει τότε ότι πρέπει να υπάρξει προσοχή, διότι μπορεί να ξεκινήσουν συγκρούσεις και να έχουμε τα ικτρά αποτελέσματα του παρελθόντος. Ένα εμφύλιο πόλεμο από το 1993 μέχρι το 2005 με 300.000 νεκρούς. Αλλά βλέπουμε πλέον ότι ο απερχόμενος πρόεδρος, ο Πιέρ Ενκουρουτζίζα, αποφάσισε να διεκδικήσει και τρίτη θητεία. Αυτό δημιούργησε αντιθέσεις, είχαμε αντιδράσεις και βεβαίως είδαμε βίαιη καταστολή. Είδαμε πάρα πολλούς να συλλαμβάνονται, έχουμε ακόμη και νεκρούς οι διώξει λοιπόν αυτέ πρέπει να σταματήσουν ο περιορισμό τη ελευθερία του τύπου πρέπει να σταματήσει. Κυρίω μα απασχολεί το πρόβλημα διότι έχουμε είκοσι χιλιάδες πρόσφυγες οι οποίοι για να γλιτώσουν πηγαίνουν στη ρουάντα και στη λαϊκή δημοκρατία του κονγκό. με τον κόδωνα του κινδύνου διότι μπορεί να έχουμε τεράστια προσφυγικά κύματα από τη χώρα αυτή και ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα. ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό τώρα ο συνάδελφος Ιβαν Γιάκοψιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι αντιμετωπίζουμε αυτό τον καιρό τώρα ένα νέο πόλεμο. Είμαστε στα πρόθυρα ενός νέου πολέμου συγκεκριμένα. Υπάρχει κίνδυνος κρίσης και ανάφλεξης και ε, μαζικής ε, αποχώρησης προσφύγων που ήδη έχουν αρχίσει. Και τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ε, πληρώσει το μερίδιο που της αναλογεί σε μια κρίση ε, που προκάλεσαν κάποιοι φίλοι της Ευρώπης και μάλιστα και η ίδια Ευρώπη, ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Θα πρέπει να δράσουμε για να μην ε, ε, ξεσπάσει αύριο ε, κρίση στη γειτονιά μας. Τα όσα βλέπουμε στη Μεσόγειο είναι αποτελέσματα αδράνειας και ολιγορίας γιατί δεν δράσαμε εγκαίρω σε κάποιες χώρες της Κεντρικής Αφρικής. Ιδού σήμερα μπροστά μας το Μπουρούντι. Το μήνυμα λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κομισιόν θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Ζητούμε στο Μπουρούντι να ε, μην ε, γίνονται τέτοια έκτροπα και από προσωπικότητες που δεν χαίρουν εκτίμηση και υποστήριξη. Ευχαριστώ πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Μίμητσα, κύριο Σκαστάλτο, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δυστυχώς ξαναμιλάμε για νιωστή φορά για τον Μπουρούντι και πρέπει να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει μια δημοκρατική ρήξη και των συμφωνιών σε του 2000. Ο σημερινός Πρόεδρος αντισυνταγματικά θέτει υποψηφιότητα ε, και νομίζω ότι αυτή η υποψηφιότητα δηλώνει την ε, συνολική έλλειψη υπευθυνότητα στην πολιτική αλλά και προστασίας της ευημερία του λαού. Αγγυλώνεται ε, στην εξουσία ε, αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες όπως ε, και το ότι πολλοί πολίτες διέφυγαν προς τις όμορες χώρες μας κάνουν να καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι ως Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσουμε κάθε τη στάση και να σκίσουμε κάθε δυνατή πίεση για να καταλάβει ο Πρόεδρος ότι δεν είναι κατάλληλη αυτή η υποψηφιότητα και θα μπορούσε να ξανακάνει τη χώρα να βουλιάξει στην γενοκτονία και στον εμφύλιο πόλεμο. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να προλάβουμε μια καταστροφή πριν να λάβει χώρα και ελπίζουμε ελπίζουμε ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να το εμποδίσουμε αυτό. Thank you very much. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα επανερχόμαστε για να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το λόγο έχει ο Επίτροπος κ. Μίμητσα. Παρακαλώ. Thank you, President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, εξωτερικό μέλη του Κοινοβουλίου. Ήταν χρήσιμη νομίζω η ανταλλαγή απόψεων που είχαμε και θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σαφήνεια με την οποία εκφραστήκατε. Όσον αφορά τώρα την αποστολή παρατηρητών και τον συντονισμό των εκλογών, πρέπει να σας πω ότι έχουμε συνεργαστεί με τους προσώπους μας επιτόπου ε, και με την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών, η οποία επίσης θα στείλει παρατηρητές και της Αφρικανικής Ένωσης και εκείνους τους ε, παρατηρητές εκλογών. Προσπαθούμε να συντονιστούμε και οι τρεις οργανισμοί μαζί. Από την συζήτηση που είχαμε, ε, αντλώ τρία συμπεράσματα. Πρώτον, ότι μας υποστηρίζει το Κοινοβούλιο στην προσπάθειά μας να εξετάσουμε όλα τα ενδεχόμενα και όλα τις δυνατότητες που έχουμε στην, ε, στα χέρια μας με βάση τη Συμφωνία του Κοτονού, εάν δεν ε, βρεθεί κάποια λύση. Ιδιαίτερα όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και Μελιωδών ελευθεριών. Δεύτερον, ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε το λαό του Μπουρούντι που βρίσκεται ήδη σε μια ευαίσθητη περιοχή και χώρα από ακόμα περισσότερε δυσκολίε όσον αφορά την οικονομική του κατάσταση και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και τρίτον, είμαστε... θέλουμε να υποστηρίξουμε τι εκλογέ με όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μα και πρέπει να εξηγήσουμε με σαφήνεια στι αρχέ του Μπουρούντι τι σημαίνει ελεύθερε εκλογέ για εμά και να παρακολουθήσουμε ε, το τι θα συμβεί, τις εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Ε, είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε, συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση και υπογραμμίζω τη σημασία που έχει ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε αυτό το θέμα να τίθεται στη Διεθνή ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε.